Ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση για τη Λευκορωσία, αγαπητοί συνάδελφοι, και μπορούμε να περάσουμε στι ψηφοφορίε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν καταρχά έξι προτάσει ψηφίσματο για τη Σρι Λάνκα. Μετά την έκθεση των ε, Ηνωμένων Εθνών, την παρακολούθηση της έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Από ό,τι έχω καταλάβει, ο κύριο Μαρέ θέλει να καταθέσει μια προφορική τροπολογία. Πρόεδρε, Εκ μέρου τη κυρία Ντεκάιζερ, καλούμε την είπατε εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο να στηρίξουν περαιτέρω προσπάθειε ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία λογοδοσία στη Σιλάνκα και να ε, εγκρίνουν την έκθεση του ΙΕ. Ιδίω την άμεση ίδρυση ενό μηχανισμού, διεθνού μηχανισμού δικαιοσύνη, απόδοση δικαιοσύνη. Υπάρχουν αντιρρήσει, κύριε Φανόρντεν. Πρόεδρε, είχαμε πολύ εντατικέ διαπραγματεύσει μεταξύ έξι πολιτικών ομάδων για αυτό το ψήφισμα. Ε, είναι συμβιβαστική λύση έτσι κι το ψήφισμα στο σύνολό του και περιέχει πολλά στοιχεία ε, για τα οποία πολλοί από εμά δεν συμφωνούσαμε. Και πολλά δεν τα συμπεριλαμβάνει. Στοιχεία τα οποία κάποιοι από εμά τα επιθυμούσαμε ιδιαίτερα. Η συμφωνία λοιπόν μεταξύ των έξι πολιτικών ομάδων ήταν να μην υπάρξουν περαιτέρω τροπολογίε πέραν των γραπτών είτε γραπτέ μάλιστα, είτε οποιασδήποτε άλλη μορφή. Είναι παραβίαση των όσων συμφωνήσαμε. Θα ήταν ε, κενέ νοήματο η διαπραγματεύσει, εάν τώρα υποβάλλεται έτσι μια τροπολογία. Εγώ λοιπόν πρέπει να την απορρίψω. Και νομίζω ότι πρέπει να την απορρίψουμε όλοι. Okay. Μάλιστα. Ποιοι λοιπόν διαφωνείτε, αν μπορείτε να σταθείτε όρθιοι για να δούμε πόσοι διαφωνούν. Yeah. than, than Νομίζω ότι είναι περισσότεροι από 10, είστε περισσότεροι από αρκετοί. Ψηφίζουμε.